Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσει σχετικά. Όχι. Οπότε θεωρούνται εγκεκριμένα τα συνοπτικά πρακτικά. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακολουθεί η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο για βιώσιμες επενδύσεις, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και Χάρτης Πορείας για την Κοινωνική Ευρώπη. Θυμίζω ότι αν θέλετε να λάβετε το λόγο στη διαδικασία γαλάζια κάρτα ή κατσιάι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο ή την ηλεκτρονική. Στην είσοδο του ημικυκλίου έχετε τι σχετικέ οδηγίε. Θα δώσω μέσα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριο Φρανς Τίμερμανς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη, μόλι τον περασμένο μήνα, δέκα μέρες αφού το ανέλαβε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τη νέα πράσινη συμφωνία. Απάντηση σε εκατομμύρια πολιτών που ζητούν ένα χάρτη έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να είναι ε, η πρώτη ήπειρο στο μπλοκ ε, που το 2050 θα είναι ουδέτερη ως προς το δεξίδι του άνθρακα και λίγες μέρες αργότερα ήρθαμε να κάνουμε την οικονομική πρόταση για ε, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης που είναι μια υπόσχεση για αλληλεγγύη και δικαιοσύνη ε, για εκείνους που ε, έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτή την κοινή μας πορεία. Θα σας μιλήσω για τις επενδύσεις στη συνέχεια, αλλά αρχίσω από το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, αν μου επιτρέπετε. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι ένα μήνυμα ε, προς τη Δυτική Μακεδονία, τους ανθρακορίχους εκεί, ε, την ε, Ισπανία και την Πολωνία, καθώς επίσης και εκείνους που εξαρτώνται από την Τύρφη στην Ιρλανδία και σε άλλες περιοχές. Ξέρουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα και η προοπτική για ένα πιο καθαρό μέλλον μπορεί να είναι γενικά ευπρόσδεκτη, αλλά ο δρόμος ε, σήμερα προς τα εκεί μας φαίνεται απειλητικός. Αυτός ο μηχανισμός για τη δίκαιη μετάβαση με 100 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μια υπόσχεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό σας σε αυτή την περίοδο, τη μεταβατική. Τρεις πυλώνες προτείνουμε για να γίνει αυτό. 7,5 δισεκατομμύρια φρέσκο καινούριο ευρωπαϊκό χρήμα, εκτός από τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το μελλοντικό προπολογισμό τη Ένωση, το Ταμείο δίκαιε μετάβαση. Αυτό θα φέρει 30 με 50 δισεκατομμύρια επενδύσεων. Χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζομένοι για μετεκπαίδευση στα επαγγέλματα του μέλλοντο, υποστήριξη στι επιχειρήσεις για νέε ευκαιρίε επένδυση σε καθαρή ενέργεια και μετασχηματισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για να προετοιμαστούν για τις νέες δραστηριότητε. Δεύτερον, Invest EU είναι το επενδυτικό μας πρόγραμμα και θα αφιερώσουμε ιδιαίτερο κεφάλαιο εκεί στη δίκαιη μετάβαση με ιδιωτικά κεφάλαια που θα φτάσουν τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να έρθουν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις και βιομηχανίες για να αντικαταστήσουν τις ρηπογόνες. Όπου θέλουν ε, οι εταιρείε να προχωρήσουν προ την ουδετερότητα, προ το κλίμα. Θα του βοηθήσουμε με νέε τεχνολογίε και για τη διατήρηση ε, θέσεων εργασία. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα υποστηρίξουν οικονομικά δημόσιου ε, φορεί, οργανισμούς, περιφέρειες, δήμους και κοινότητε, για προγράμματα που θα βοηθήσουν ας πούμε, τον κόσμο να μονώνει τα κτίρια. Με σύγχρονα συστήματα θέρμανση για οικογένειε που ακόμα εξαρτώνται το χειμώνα για να ζεσταθούν από τον άνθρακα ή το ξύλο. Ξέρουμε ότι οι ε, περιοχές που πλήττονται περισσότερο χρειάζονται ειδική στήριξη γιατί ψάχνουν εναλλακτικέ λύσεις. Όλες οι περιφερειακές λοιπόν εμπειρίες θα συνενωθούν σε αυτή την πλατφόρμα δικής μετάβασης. Η σημερινή μας πρόταση είναι κατεπίγουσα. Το Κοινοβούλιο το γνωρίζει καθώς ε, ε, έχει την πλατφορμα δική μετάβαση. η σημερινη μας προταση ειναι επιγουσα ιδιοκτησία αυτής της υπόθεσης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ελπίζουμε και περιμένουμε το, κοινοβούλιο, να το, το Συμβούλιο συγγνώμη, γρήγορα να το εγκρίνει και να το ετάξει στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιε είναι οι περιοχές που χρειάζονται τα χρήματα και την πρακτική μας υποστήριξη και να εργαστούν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι συλλογική αυτή η προσπάθεια. ΟΤΑ, κοινωνικοί εταίροι, βιομηχανίες, κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συνεργαστούν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και την ιδιοκτησία θα πρέπει να την έχει η περιφέρεια και οι πολίτες να το υποστηρίξουν. Ξέρουμε ότι αυτά τα 100 δις είναι αρχή και μόνο. Η δικαιοσύνη ξεπερνάει κατά πολύ αυτό το μηχανισμό. Η ε, κλιματική αλλαγή θέτει νέα θεμέλια στην ε, κοινωνία μας. Χρειαζόμαστε καθαρό αέρα, καθαρό νερό και ε, οι πιο ευάλωτοι θα πρέπει να επωφελούνται. Η δικαιοσύνη είναι πάντα στο μυαλό μας ε, θέλουμε ε, να είναι ε, το περιβάλλον και το μέλλον καθαρό αλλά και βιώσιμο και προσιτό. 400.000 πρόωρους θανάτους έχουμε στις πόλεις μας από τα καυσαέρια, τα δελτηριώδη που αναπνέουν οι πολίτες. Έχουμε τις δυνατότητες, τα μυαλά και τη τεχνολογία να φέρουμε αποτελέσματα στην Πράσινη Συμφωνία. Σήμερα αναλαμβάνουμε αυτή την υποχρέωση και όχι μόνο αυτή, δεν θα αφήσουμε κανέναν ε, πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει αντιπρόεδρος κύριος Βάλτης Δομπρόφσκης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει τις φιλοδοξία μας, τη φιλοδοξία μας ε, ε, να γίνει μέχρι το 2050 η Ευρώπη ουδέτερη σε ό,τι αφορά τον άνθρακα. είναι κάτι που οφείλουμε στους πολίτες μας και σε επόμενες γενιές. Πρέπει να πετύχουμε το πρόγραμμα βιώσιμων επενδύσεων ή το πρόγραμμα που θα στηρίζει τη Νέα Πράσινη Συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα από την Κομισιόν ε, υλοποιεί αυτή, αυτή ακριβώς τη φιλοδοξία και προβλέπει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Ε, προβλέπει ε, καινούργιες νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες αλλά τη συνδέει και με υπάρχοντα ε, ταμεία και εργαλεία. Να σας υπογραμμίσω τους τρεις πυλώνες μας. Πρώτον, χρηματοδότηση. Θα κινητοποιήσει το σχέδιο αυτό τουλάχιστον ένα 3 ευρώ ε, βιώσιμων επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει το μισό από αυτό το ποσό και θα χρησιμοποιήσουμε και μόχλευση. Το Invest EU θα κινητοποιήσει περίπου 279 δισεκατομμύρια ευρώ από κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση ε, με περιβαλλοντικές επενδύσεις ε, και θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο εμείς το παράδειγμα. Η Εθνική Συγχρηματοδότηση Οικολογικών Σχεδίων θα φέρει επίσης 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης ε, θα είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο πολιτές μεσονικό πλαίσιο. Επίσης, έχουμε το <clears throat> το Ταμείο Καινοτομία και τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ η οποία θα περάσει από το 25% στο 50% μέχρι το 2025. Ε, επίσης, θα επιτρέψουμε